Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισε την οδηγία γιατί δεν είναι σωστός συμβιβασμός μεταξύ των δικαιωμάτων των δημιουργών και των χρηστών. Θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί άλλες λύσεις. Αλλά ειδικά οι κάτοχοι των δικαιωμάτων και η πλειοψηφία εδώ του Κοινοβουλίου δεν βλέπει ε, επαρκώς τον κίνδυνο που υπάρχει στα φίλτρα ανεβάσματος και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό λάθος. Οι παραγωγοί περιεχομένου θα διαπιστώσουν ότι θα εισπράξουν λιγότερα από όσα ελπίζουν. Θα προωθηθεί ένα μονοπόλιο ισχύω στο διαδίκτυο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι πραγματικά απογοητεύονται από αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Σας ευχαριστώ. Χάρκιν. Ήταν μια καλή ημέρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε τα δικαιώματα δημιουργών, καλλιτεχνών και λοιπόν για μια δίκαιη ανταμοιβή για την εργασία τους. Αυτό το κάναμε με το να υπάρχει προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας όταν χρησιμοποιείται αυτή για κέρδος από ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι μια νίκη για τα άτομα καθώς οι πλατφόρμες πλέον δεν θα μπορούν να συσσωρεύουν τεράστιες ε, περιουσίες στην πλάτη των δημιουργών με την εκμετάλλευση του έργου τους. Σήμερα το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να υποκύψει στις καμπάνιες αυτών που θέλουν να διατηρήσουν την κυρίαρχη θέση τους. Και τέλος, μία από τις αρχές στις οποίες πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αρχή της αξιοπρεπούς πληρωμής για τους εργαζόμενους και για τον κόπο τους. Νομίζω λοιπόν ότι τηρήθηκε σήμερα αυτή η αρχή για τους δημιουργούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ομαρζή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ προστασία των δημιουργών και η αντίσταση στις μεγάλες πλατφόρμες δεν σημαίνει ότι αντιτιθέμεθα ε, στις μικρές πλατφόρμες και κατά της νομοδότησης ε, της τάσης του ΟΗΕ ούτε κατά των πανεπιστημίων, ούτε κατά των εκατομμυρίων πολιτών ε, στην Ευρώπη που ε, προβληματίζονται και ανησυχούν ε, για την ποιότητα της πληροφορίας, γιατί η ελευθερία της έκφρασης και η ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων απειλούνται από το μαζικό φιλτράρισμα του περιεχομένου, το οποίο προετοιμάζεται με αυτή την οδηγία. Ένα κείμενο το οποίο θεωρώ επιζήμιο προς την ελευθερία. Αυτή η οδηγία είναι παροχημένη και διαβρώνεται από μία αντίληψη του διαδικτύου του προηγούμενου αιώνα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο διαδίκτυο που πραγματικά θα προστατεύει ε, το περιεχόμενο και θα φορολογεί πραγματικά τους μεγάλους. Ο κύριος Κέλλιν. Ευχαριστώ. Το απλούστερο σήμερα θα ήταν να απόσχουμε ή ε, να κάνουμε ότι δεν είμαστε εδώ και να μην ψηφίσουμε καθόλου. Αλλά αυτό δεν είναι η δική μου πεποίθηση. Πάντα ψηφίζω και υπερψήφισα αυτή την αμφιλεγόμενη αλλά σημαντική πρόταση. Κατανοώ τους προβληματισμού που ετέθησαν. Πρέπει η νομοθεσία να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξει αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία τη αστική αγορά στηρίζω την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων από τις παραβιάσεις. Πρέπει να υπάρχει δίκαιη ανταμοιβή προς τους δημιουργούς και να βρεθεί και μια σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων τους και αυτών των οικονομικών ψηφιακών φορέων. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Αντί όλα τα έσοδα να πηγαίνουν μόνο στις τσέπες των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Η ψηφιακή εσωτερική αγορά δεν είναι μόνο οικονομικό φόρουμ, αλλά και πολιτιστικό. Κανένας φορέας, κανένας δημοσιογράφος θα πρέπει να βλέπει το έργο του να ε, την χάνει εκμετάλλευση χωρίς αυτός να λαμβάνει καμία ανταμοιβή. Μπορεί να βελτιωθεί βέβαια η πρόταση σε ό,τι αφορά την υλοποίησή τη σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ, Σκύρπεκ. Ευχαριστώ πολύ. Στην eh, ψηφιακή εποχή θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι συντάκτες της οδηγίας έχουν αποτύχει. Επειδή ακριβώς ε, θέλω, ε, καταψήφισα, ε, ε θλίβαμε για το γεγονός ότι οι πολίτες ε, τάχθηκαν υπέρ. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη συνιστούν σημαντική πρόκληση για τη δημοκρατία και παρέχουν σε αυταρχικούς ε, ηγέτες ε, νέα προπαγανδιστικά μέσα. Ε, και τα νέα έργα είναι, τα νέα αυτά προϊόντα είναι άκρος επικίνδυνα. Εγώ ο ίδιος είμαι μεταφραστής πολλών βιβλίων οι εκδότες και οι δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να βλέπουν τα... Ε, θα πρέπει να έχουν μια εγγύηση των πνευματικών τους ε, δικαιωμάτων. Υπάρχει ανθολικές χώρες πλούσια εμπειρία όσον αφορά τις ε, προσπάθειες περιστολής των ελευθεριών. Η κυρία Λέρνερ. Σας ευχαριστώ. Πολλές ΜΚΟ και πολλοί εμπεριγνώμονες εδώ άσκησαν ε, ισχυρή κριτική, έντονη κριτική σε αυτή τη νέα οδηγία. Εγώ ανησυχώ σε σχέση με το αυτόματο φιλτράρισμα των κατεβασμάτων και σχετικά με τους αλγόριθμους Μπορεί να υπάρξει δηλαδή αυτόματη λογοκρισία και να υπάρχει περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης των πολιτών στο διαδίκτυο. Οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις έχουν μικρότερες δυνατότητες ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνισμού. Η οδηγία επίσης ε, αλλάζει τη λογική των συνδέσμων για τις ειδήσει και τον όγκο των ειδήσεων. Ε, κερδίζουν οι μεγάλοι, χάνουν οι μικροί. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύεται το δικαίωμα του δημιουργού στο διαδίκτυο. Θα πρέπει οι δημοσιογράφοι επίση ε, να αμείβονται. Ο κίνδυν, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή τη μεταρρύθμιση είναι τεράστιοι. Γι' αυτό καταψήφισε αυτή την πρόταση και κυρίω κατά των άρθρων που είναι προβληματικά. Σα ευχαριστώ, ο κύριο Σουσνιέρ. Ναι, εγώ είπα ότι δεν θα έπρεπε να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πραγματικά μας μεταχειρίζεται με το μαστίγιο. Τώρα δεν έχουμε μόνο το μαστίγιο λοιπόν της Βαρσοβίας, αλλά έχουμε και το δεύτερο μαστίγιο των Βρυξελών. Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της μαστίγωσης των Βρυξελών ε, και της Βαρσοβίας. Ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, δεν έχουμε καμία καλή πρόσβαση στον ε, πολιτισμό, οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων δεν ε, έχουν ε, την απαραίτητη εγγύηση των έργων τους. Όχι. Όλα αυτά συνιστούν πρόσχημα προκειμένου να ελεγχθεί το τελευταίο προπήγιο των φιλελεύθερων αξιών στην Ευρώπη. Το διαδίκτυο είναι μια απόδειξη ότι ο κόσμος μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ε, ανώτιτους περιορισμούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως ο απλούστερος ε, τρόπος να απαντήσουμε σε μια τέτοια ψηφοφορία θα ήταν να απόσχουμε, λέει ο κύριος Πόλτσακ. Αλλά αυτό δεν επαρκεί. Θεωρώ ότι οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων, είτε είναι ε, ιδιοκτήτε των λογισμικών, είτε δημιουργοί, ε, πρέπει να ανταμείβονται για το περιεχόμενό τους. Και φυσικά και οι χρήστες από την άλλη πρέπει να είναι σε θέση ε, να έχουν συγκεκριμένους όρους για την χρήση των αδειών. Τελικά μας απογοητεύει το σημερινό αποτέλεσμα γιατί δεν καταφέραμε να ψηφίσουμε επιτροπολιγιών. Για το άρθρο 13 ήταν αυτό. Το, το 11 ήταν ισορπημένο. Το 13 όμως άλλαξε στον τριμερή διάλογο και τώρα πλέον ε, είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Θα πρέπει να διορθωθεί αυτό. Δεν ε, καταφέραμε να το κάνουμε αυτό σήμερα εξαιτία τη διαδικασία ε, που ακολουθήθηκε, γι' αυτό και τελικά απήχα. Ευχαριστώ κύριε Μαμίκινς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορώ να συγχαρώ εμάς και τους συναδέλφους μας ε, γιατί ψήφισαμε υπέρ μιας λογοκρισίας στο διαδίκτυο. Και δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι χειροκρότησαν τον κύριο Φως όταν ε, έγινε αποδεκτή και αυτή η προσθήκη. Εγώ Ήμουν υπέρ της πρότασης της κυρίας Ρέγκνερ να υπάρξουν τροπολογίες και καταψήφισα την πρώτη ανάγνωση. Όμως πραγματικά να σας συγχαρώ. Πηγαίνουμε στην ε, κατεύθυνση της Βόρειας Κορέας και της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Και οι συγγραφείς δεν θα λαμβάνουν τίποτα γιατί οι μεγάλες εταιρείες ε, θα παίρνουν τα χρήματα. Στη λετωνική τηλεόραση Είχαμε έναν κωδικό μετάδοσης χωρίς λογοκρισία, όμως τώρα θα υπάρχει λογοκρισία. Εμείς στην Ανατολική Ευρώπη τα καταλογούμε πολύ καλά αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει λογοκρισία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόταση ψηφίσματο για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανική καταγωγή, η κυρία Κίνγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για πρώτη φορά η Ευρώπη αναγνωρίζει αυτή την μισητή μορφή ρατσισμού απέναντι στα άτομα αφρικανικής καταγωγής. Δυστυχώς γιατί δεν το λένε και πιο πολύ στην Ευρώπη. Αυτό το ψήφισμα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα προς μια κοινωνία πολυπολιτισμική, ισότιμη και όπου θα υπάρχει σεβασμός. Μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει πλέον χώρος για το ρατσιστικό μίσος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη έκθεση. Κόφορτ, ε, Νίντερ Μάγερ, για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροποφυγή. Η κυρία Μακοβέ έχει το λόγο. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με εξοστίζει 110 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει το 1% του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, το 70% των περιπτώσεων της ε, ξεπλήματος χρημάτων είναι διασυνοριακές. Σε παγκόσμιο επίπεδο το κόστος φτάνει για από πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πέρσι υιοθέτησαν την πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση τη νομοποίηση παράνομων εσόδων. Υπάρχει λοιπόν νομοθετικό πλαίσιο τη Ένωση για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου και θα πρέπει να μεταφερθεί στο ιστορικό δικαίο η νομοθεσία μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Ούτε την τέταρτη οδηγία δεν έχει μεταφέρει η Ρουμανία και ξεκίνησε η Κομισιόν την διαδικασία επιπεραβάση κατά της Ρουμανίας και γιατί έχει καθυστερήσει, αλλά και γιατί στη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο δεν σέβεται τι προβλέψει τη τέταρτη οδηγία. Η κυβέρνηση Ρουμανία θα πρέπει να υιοθετήσει άμεσα την οδηγία και να μεταφέρει εγκαίρω τι ευρωπαϊκέ Οδηγίε στο ιστορικό δίκαιο. Διαφορετικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνο αν όλοι σωστά μεταφέρουμε στο ιστορικό μα δίκαιο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Μάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι δίκαιο ούτε ηθικό και είναι και υπερβολικό. Η υπερβολικά πλούσια παγκόσμια ελίτ που αποφεύγει να πληρώνει το μερίδιό τη, ε, αποστέλνοντα τα χρήματά τη σε φορολογικού παραδείσου ανά τον κόσμο, θα πρέπει να παρεμποδιστεί. Όλα αυτά τα χρήματα ανήκουν στι τάξει των σχολείων μα, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά μα τμήματα. Και είναι πραγματική προσβολή και προ τους ε, απλούς φορολογουμένους που πληρώνουν ε, κανονικά το μερίδιό τους και τους φόρους τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πιέσει και να προωθήσει ε, πραγματικέ μεταρρυθμίσει. Γι' αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να σταθεί σε αντίστοιχο ύψο, είτε επέλθει το Brexit είτε όχι. Και δεν θα πρέπει να υπάρξει μία, ε, ένας αγώνας προς τα κάτω σε ό,τι τη φορολογία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πέντε χρόνια σε ειδικέ επιτροπέ συνεργάστηκα τα κείμενα 1, 2, 3 για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, αλλά και στην Εξωτική Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά. Έλαβα μέρο σε πολλέ ακροάσει με υπουργού οικονομικών, τραπεζίτε κλπ. Το έργο πολλών δημοσιογράφων αλλά και καταγγελών τον άξιζε τον κόπο. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω και στην ε, Δάφνη την Καλίτσια η οποία δολοφονήθηκε. Ε, το φαινόμενο που το ξέπλυμα χρημάτων θα πρέπει να γίνει, ε, να παρεμποδιστεί. Ο αγώνας κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει να ενισχυθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, συνεχίσει αυτή την προσπάθεια και οι χώρες μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη συνεργασία τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη όσον αφορά το φορολογικό σύστημα. Ο κύριος ε, Ζηροζεύσκη αν ε, ήξερα τι θα έλεγε ο κύριος ε, Μαν, δεν θα ζητούσα το λόγο γιατί με κάλυψαν απολύτως τα λόγια μου. Ε, και εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι οι εργασίες διήρκεσαν μεν μόνο ένα χρόνο, αλλά ευθύς εξ αρχής το κοινοβουλευτικού μας, από την αρχή του κοινοβουλευτικού μας έργου καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες παρόλο που προσπάθησαν να μας βάλουν εμπόδια στο δρόμο μας. Παρόλα αυτά μπορέσαμε να επεξεργαστούμε πάρα πολλούς συμβιβασμούς και τελικά η έκθεση αυτή μπόρεσε να ε, περάσει και προλυαίνει ε, το δρόμο τον οποίο ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ροζάτη. Θα ήθελα με μεγάλη ικανοποίηση να χαιρετήσω την έγκριση αυτής της, την υπερψήφιση αυτής της έκθεσης. Η έκθεση αυτή έγινε δεκτή και χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την, μια πλατιά υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Εγώ ήμουν στο ΤΑΞ 3 και ασχολήθηκα, ε, συνεργάστηκα πολύ στενά με τους εισηγητές προκειμένου να πετύχουμε ε, το συμβαστικό αποτέλεσμα το οποίο μπόρεσε να υποστηριχθεί από το πλατή φάσμα των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτελεί το επιστέγασμα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας την οποία, της οποίας ηγήθη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αποτέλεσμα ήταν η προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλήματος των, ε, χρημάτων ε, για παράδειγμα να αποτελέσει μια σημαντική προτεραιότητα της μας. η κυρία ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή είναι πολύ εκτεταμένες. Η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή του ΦΠΑ επιφέρει σημαντικές ε, ζημίες οι φορολογικές αρχές των χωρών μελών δεν συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και η ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι ιδανική. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Πέραν τούτου, ε, ορισμένες περιφέρειες δεν είναι ιδιαίτερως αποτελεσματικές όσον αφορά τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή και δεν προτίθεται να αναλάβουν αυτή την προσπάθεια. Ε, μικρές ε, επιχειρήσεις αναγκάζονται να πληρώνουν ακριβούς φορολογικούς συμβούλους. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, υφιστάμενες ε, διατάξεις. Αυτό θα είναι πολύ θετικό για την πολιτική των χωρών μελών. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εφόσον θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Στη σημερινή ψηφοφορία εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπεθ, η κυρία Λόπεθ Βερμέχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η φοροδιαφυγή και η υποφυγή είναι ένα θέμα που προσκάπτει τις οικονομίες μας, αφαιρεί πόρους που μπορούσαν, θα μπορούσαν να δοθούν για την ευημερία των πολιτών ε, και μειώνει την εμπιστοσύνη στους ε, θεσμούς. Το ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν είναι ίδιες για όλους έχει αυξήσει τη σύγχυση και την οργή στις κοινωνίες μας. Δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι η φορολογική ποιήση και απαιτήσει ε, πάντοτε είναι για το λαό και για τις μεσαίες τάξεις. Η αποφορολόγηση των εισοδημάτων επίση σήμαινε σοβαρή επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες στις πόλες στις χώρες μας ε, υπό τη δικαιολογία ότι με λιγότερους φόρους ε, πρημοδοτείται η απασχόληση. Οδηγηθήκαμε στη φτώχυνση των κρατών ε, και δυσκόλεψαν οι κοινωνικές πολιτικές. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί η Επιτροπή Tax 3 εργάστηκε καλά και αποκάλυψε μέχρι ποιο σημείο οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μηχανισμούς φορολογικού σχεδιασμού όλο ένα και πιο επιθετικού για να μη σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Η ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων είναι η μεγάλη τρύπα που επιτρέπει τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή από την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων και των εχόντων. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η διαφορετικότητα των φορολογικών μοντέλων στην Ευρώπη δημιουργεί έναν ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών που τον εκμεταλλεύονται οι μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να συνεισφέρουν όλο ένα και, και λιγότερο. Σε αυτή την ανταγωνιστική λογική, κανένα δεν κερδίζει και όλοι χάνουμε. Νωρίτερα ή αργότερα κάποιο μπορεί να βάλει πιο χαμηλού φόρου και να προσφέρει καλύτερα φορολογικά πλεονεκτήματα. Ο ανταγωνισμό προ λιγότερα δικαιώματα ζημιώνει τη μεγάλη πλειοψηφία. Γι' αυτό τώρα ε, πρέπει να υπάρξει ένα συμβιβασμό των χωρών για να εφαρμοστούν οι διατάξει τη πρόταση, αν πραγματικά θέλουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και θέλουμε να μειωθεί η κοινωνική οργή. Τότε θα πρέπει να εγγυηθούμε τα ελάχιστα έτσι ώστε οι κοινωνίε μα να εμπιστεύονται τους θεσμούς τους. Και το φορολογικό σύντημα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό για την υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Διακόπτουμε τώρα μέχρι τις 3. Σας ευχαριστώ.